και σας ευχαριστούμε επίσης για όλη την βοήθεια και τη συνεργασία που είχαμε μαζί σας. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα που είναι η εμπορία ανθρώπων. Πρώτος ομιλητής η κυρία Αναχέντ για δυόμιση λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρουμε όλοι, η εμπορία ανθρώπων είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα στον κόσμο, γι' αυτό και είναι πραγματικά κρίμα που τόσο αργά και σε μια σχεδόν άδεια αίθουσα και χωρίς ε, κανένα δημοσιογράφο αποφασίζουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Έχει εγκαταλειφθεί και καταργηθεί η δουλεία πριν από... 150 χρόνια, το 1850. Βλέπουμε όμως ότι συνεχίζει μια παρόμοια μορφή εκμετάλλευσης και δουλείας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεράστια ευθύνη και θα πρέπει εδώ να καταπολεμήσουν αυτήν την δουλεία σεξουαλική είτε εργασία υποχρεωτική και καταναγκαστική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν στην προετοιμασία αυτού του κειμένου και ελπίζω όλοι μαζί να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Ελπίζω επίσης η νέα Επιτροπή να αναλάβει την προετοιμασία μιας νέας οδηγίας η οποία θα αντικαταστήσει την παλιά πρόταση. Ένα κείμενο που δεν ήταν κακό, αλλά ίσως θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη προοπτική σήμερα στις προτάσεις μας, μια πρόταση η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το ποινικό τμήμα αυτής αυτού του φαινομένου, αλλά και το θέμα της μετανάστευσης, ένα φαινόμενο που επιδεινώνει την κατάσταση. Επίσης θα πρέπει να επιμείνουμε στις ε, απτές συνέπειες αυτού του φαινομένου, τις κυρώσεις και ιδιαίτερη προστασία για τα ανήλικα θύματα. Χρειάζεται συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Την ίδια ώρα, πολύ σημαντική είναι και η πρόληψη τη εμπορία ανθρώπων. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν και να καταπολεμήσουν και την ζήτηση. Εάν η ζήτηση καταπολεμηθεί, τότε το φαινόμενο θα υποχωρήσει. Σε αυτή την περίπτωση η προσφορά θα μειωθεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να στραφώ προς το σύνολο των θεσμικών οργάνων, προς τα κράτη-μέλη και να ζητήσω από όλους να συντονίσουμε τη δράση μας έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε αυτήν την σύγχρονη δουλεία που είναι η εμπειρία των ανθρώπων. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπάουερ για μισή λεπτά έχει το λόγο. Η εμπορία ανθρώπων είναι σοβαρότατο θέμα εκατοντάδες χιλιάδες άτομα σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι θύματα αυτής της εμπορίας. Είναι κάτι το απίστευτο, απίστευτο. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι αυτό είναι οριακό φαινόμενο, του οποίου τη σημασία υποτιμούν. αλλά δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα και γι' αυτό το λόγο η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Θα μιλήσω για δύο θέματα. Πρώτον, προστασία των θυμάτων και δεύτερον, μείωση της ζήτησης. Παρόλο που υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των θυμάτων και η Επιτροπή υποσχέθηκε να την ξαναδεί, να την επαναξιολογήσει αυτή τη νομοθεσία το 2009 μιλάμε για ένα νομοθετικό κείμενο του 2004 που πρόκειται να αναθεωρηθεί ώστε να αναβαθμιστεί η προστασία των θυμάτων. Διότι χωρίς μια τέτοια προστασία δεν θα μπορέσουμε να εξαρθρώσουμε τις σπήρες του οργανωμένου εγκλήματος. Και Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο θέμα της δημιουργίας ζήτησης, διότι υπάρχει μια αγορά για το εμπόριο ανθρώπων. Και αυτή η αγορά στηρίζεται στους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, όπως και όλες οι υπόλοιπες αγορές. Έχουμε την τάση να αγνοούμε την πλευρά της ζήτησης της αγοράς. Έως ότου καταφέρουμε να περιορίσουμε τη ζήτηση, δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την εμπορία ανθρώπων. Και θέλω να υπογραμμίσω επίσης το γεγονός ότι απαιτείται συντονισμός των πολιτικών που χαράσουμε και εφαρμόζουμε. Οι γενικές διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσοι λαμβάνουν αποφάσεις δεν συντονίζουν τις πολιτικές τους και υπάρχει δυσχέρεια στην επικοινωνία και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Τώρα, ο κ. Λόπες Γκαρίδη για το Συμβούλιο. Επόμενος ομιλητή. Κυρίες Χέντ και Μπάουερ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την πρωτοβουλία, την ερώτηση και τη συζήτηση την οποία ζητήσατε εδώ απόψε. Νομίζω ότι η εμπορία ανθρώπων είναι το μεγαλύτερο πλήγμα της κοινωνίας και είναι και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε από κοινού. Ένα ακόμα παράδειγμα της μεγάλης σημασίας ε, το ε, να αντιμετωπίσουμε από κοινού κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πολύ πέρα από το ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πληγή. Μιλάτε για τα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσεγγίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρεστε στον επαναπατρισμό, κοινωνική ενσωμάτωση, κοινωνικά θέματα. Η απάντηση είναι ναι. Αυτό είναι ο σωστό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε και την αναλογικότητα των ποινών. Αυτό το θέτετε και εσεί στην ερώτησή σα. Και ταυτόχρονα να δούμε και κατά πόσο είναι απαραίτητα επιπλέον μέτρα για την προστασία των θυμάτων το ε, επισημάνατε και επιμείνατε και συμφωνώ απόλυτα, η προστασία των θυμάτων είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την εμπορία των ανθρώπων. Και το να μπορέσουμε να σώσουμε κάποιον ο οποίος είναι θύμα σε κατάσταση άμυνας και ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι θύμα της εμπορίας είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την εκμετάλλευση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό που μας λέτε για το θέμα της ζήτησης. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να κάνουμε ό,τι γίνεται και με το θέμα της ε, δικαιοδοσίας. Στη δεύτερη παράγραφος της ερώτησης μας φέρεται απαραίτητο να γίνει συντονισμός των πληροφοριών. Συμφωνούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την προσήγηση που προτείνει αυτή η ερώτηση και μιλάτε επίσης και για προληπτικά μέτρα. Ε, να πω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται αυτά τα ε, μέτρα πρόληψης. Ήδη από το 2005 το Συμβούλιο ενέκρινε ένα σχετικό σχέδιο, το οποίο φυσικά θα πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Και όπως γνωρίζετε, το θέμα της εμπορίας ανθρώπων περιλαμβάνεται σε πολλές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεων και τρίτων χωρών. Για παράδειγμα, τη στρατηγική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης-Εφρικής καθώς επίσης και πολλές συμφωνίες σταθεροποίησης ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική η συνδρομή στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Θα πρέπει να υπάρχει και κατάρτιση και ευαισθητοποίηση ανθρώπων που είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή με θύματα. Για παράδειγμα, ε, συνοριοφύλακες, ε, άτομα τα οποία παρέχουν βοήθεια σε τρίτες χώρες. Η Ισπανική Προεδρία και να ολοκληρώσω με αυτό, θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση, θα ασχοληθεί κυρίως με το θέμα των παιδιών, τα οποία πλήττονται από την εμπορία και αυτό είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας και ε, μεταξύ των όλων πρωτοβολιών έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει στις αρχές του 2010 ένα πρόγραμμα δράσης για τους ανήλικους που δεν συνοδεύονται και φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν κατακλείδη κύριε Πρόεδρε, η Ισπανική Προεδρία θέλει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας της να υπάρξει μια συζήτηση για μια οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και είμαι πεπισμένος ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει αμέσως μια τέτοια πρόταση. Αυτή τη στιγμή υπάρξει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ισπανική Προεδρία θα ξεκινήσει τη συζητήση στο Συμβούλιο από κοινού με το Κοινοβούλιο. Αυτό νομίζω ότι εκφράζει την αποφασιστικότητά μας και τη διάθεσή μας να καταπολεμήσουμε αυτό το σύγχρονο δουλεμπόριο όπως πολύ ε, σωστά το όρισαν οι προλαλήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρό. Κύριε Πρόεδρε, μας εξήγησε ο Υπουργός μόλις τώρα ότι πρόκειται για μια μορφή δουλείας του ανθρώπινου εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ τις δύο εισηγήτριες, τις δύο κυρίες που έθεσαν αυτή την προφορική ερώτηση. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο σφαιρική και πολυδιάστατη προσέγγιση, η οποία θα ενσωματώσει και μια διεθνή συνεργασία με τρίτες χώρες. Αυτή ήταν και η προσέγγιση της Επιτροπής όταν έκανε την πρόταση για μια συμφωνία απόφαση πλαίσιο το 2009 το Μάρτιο. Αυτή η απόφαση πλαίσιο βασίζεται στην πρώτη του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για την καταπολέμηση του εμπορίου των ανθρώπων την ξεπερνά παρόλα αυτά. Όπως ε, είπατε κύριε Υπουργέ θα χρησιμοποιήσουμε τη νέα νομική βάση που μας επιτρέπει η Συμφωνία της Λισαβόνας έτσι το ταχύτερο δυνατόν να υποβάλουμε μια πρόταση οδηγίας που θα λάβει υπόψη όλα αυτά που ακούστηκαν πριν την θέση σε ισχύ της ε, Συνθήκης Λισαβόνας. Και ελπίζουμε ότι αυτή η νέα πρόταση οδηγίας θα είναι πολύ φιλόδοξη. Έχουμε την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει εδώ να παίξει ουσιαστικό ρόλο ότι η δέσμευσή του είναι καθοριστική για να ενισχυθεί ακόμα παραπάνω το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του εμπορίου των ανθρώπων. Θα σας ε, υποβάλω εδώ κάποια στοιχεία, προσπαθώντας να απαντήσω σε αυτή την προφωτική ερώτηση. Καταρχήν, οι κυρώσεις. Η εμπορία των ανθρώπων αποτελεί πολύ σοβαρό αδίκημα, το οποίο θα πρέπει να τιμωρείται αντίστοιχα. Οι κυρώσει πρέπει να είναι αυστηρές και εδώ θα πρέπει η σύγκληση αυτών των μέγιστων ποινών να συνεχιστεί, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλήσει μεταξύ των κρατών μελών. Από 3 έως 20 έτη. 10 έτη φυλάκισης μέχρι και ισόβια φυλάκιση όταν υπάρχουν και όταν υπάρχουν σοβαρότεροι λόγοι και επιφαρετικά στοιχεία. Τεράστιες λοιπόν αποκλήσεις απαράδεκτες και αδικαιολόγητες σε μια ευρωπαϊκή προοπτική. Στην νέα λοιπόν πρόταση οδηγίας θα προτείνουμε αυστηρότατες ποινές. Όσον αφορά την προστασία των θυμάτων και την συνδρομή, η συνδρομή και η προστασία των θυμάτων όσον αφορά την στέγη, την ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική βοήθεια, συμβούλη, ενημέρωση, υπηρεσίες διερμηνίας μετάφρασης, δικαστικής συνδρομής, όλα αυτά είναι ουσιαστικά. Και όπως επιθυμεί και η Ισπανική Προεδρία θα πρέπει να προβλέπονται ειδικά μέτρα προστασίας των ανήλικων θυμάτων, των παιδιών. Η υπεράσπιση τους παραδείγματος χάρη θα πρέπει να είναι δωρεάν για τους ανήλικους. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πρώτη έκθεσή της όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας που αναφέρεται στις άδειες παραμονής υπηκών των χωρών που είναι θύματα αυτής της εμπορίας ανθρώπων και θα δούμε μετά την δημοσίευση αυτής της έκθεσης εάν υπάρχει ανάγκη για τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα για την αποθάρρυνση, αποτροπή της ζήτησης. Προβλέπει εδώ η Επιτροπή να συμπεριλάβει μέτρα για την πρωτοβουλία των κρατών μελών. Επίσης, προτείνει να δώσει κίνητρα στα κράτη-μέλη για να υπάρξουν κυρώσεις κατά του χρήστη αυτών των σεξουαλικών υπηρεσιών όταν ο χρήστης γνωρίζει ότι πρόκειται για θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις δυνατότητες των κρατών μελών να αναλάβουν μέτρα και να προσφύγουν κατά ατόμων τα οποία συμμετέχουν σε, αυτήν την, σε αυτά τα δίκτυα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σε αυτές τις νέες μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις, στις οποίες συμμετέχουν άτομα πολλών εθνικοτήτων, με έδρα πολλές φορές ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει δίκτες έτσι ώστε να μπορούν να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να ακολουθούνται από κοινά πρότυπα, να βασιζόμαστε στα στοιχεία της Eurostat, της Europol, της Eurojust, της Frontex και της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όσον αφορά την πρόληψη τέλος, υπάρχει ένα οικονομικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση και την πρόληψη αυτής της εγκληματικότητας το 2010. Θα γίνει μια συγκεκριμένη έκκληση όσον αφορά την καταπολέμηση του εμπορίου των ανθρώπων τέλος το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις στο έγγραφο Γενικού Πρωτολισμού που υιοθέτησε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο ΖΑΗ συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι η σφαιρική, η γενική πολιτική για την καταπολέμηση του εμπορίου των ανθρώπων και όπως σας είπα και προηγουμένως η Επιτροπή θα υποβάλει ένα σχέδιο οδηγίας και χαίρομαι ιδιαίτερα και διακόγοντας την Ισπανική Προεδρία συνειδητοποίησα ότι πραγματικά θα υπάρξει μία συζήτηση με σκοπό τον εμπλουτισμό της πρότασης της Επιτροπής, η οποία φαίνεται να είναι επίκαιρη, καθότι το φαινόμενο αυτό δεν υποχωρεί, αλλά παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις στις χώρες μας. Ήρθε λοιπόν η ώρα να αντιδράσουμε με δυναμικό τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η κυρία Αντζελίλη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες Χέτ και Μπάουερ για την πρωτοβουλία τους. Η εμπορία ανθρώπων, όπως είπαν όλοι πριν από μένα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αδίκαιωμα, το οποίο συνδέεται με την παιδική εργασία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι ε, δεν έχουν καμία εδώ και εκμεταλλεύονται άτομα με τη χρήση βίας ή και με δόλο. Ορισμένες φορές υπόσχονται μία τίμια δουλειά με καλές αποδοχές και υπάρχουν και πολλές φορές και εκβιασμοί κατά των θυμάτων, κατά των οικογενειών τους και των παιδιών τους. Δυστυχώς όπως πολύ συχνά συμβαίνει οι γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά είναι αυτά τα οποία πληρώνουν το τίμημα. Εκτιμώνται ότι είναι περίπου 2 εκατομμύρια τα θύματα της εκμετάλλευσης ε, παγκοσμίω και το 80% περίπου αποτελείται από γυναίκες και παιδιά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ανηλίκων είχε καταγγείλει ότι η εμπορία παιδιών έχει πάρα πολλούς εγκληματικούς σκοπούς. Εμπορία οργάνων, ε, πορνεία, παράνομη εργασία, ε, υποχρεωτική γάμη, επαιτία. Ε, αυτά είναι για να σας δώσω κάποιο παράδειγμα. Σε αυτό το έγγραφο ε, η εμπορία θεωρήθηκε μια πραγματική πληγή και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως η καταπολέμηση της εκμετάλλευσης έπρεπε να γίνει προτεραιότητα για το μελλοντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως υιοθετώντα όλα τα νομοθετικά μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα και κατεπήγοντα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πλήρης προστασία και συνδρομή προς τα θύματα. Μιλήσαμε για εκμετάλλευση και κακομεταχείριση ανηλίκων και στο πρόσφατο πρόγραμμα της Στοχόλμης. Εν κατακλείδη λοιπόν και βάσει της απόψινής συζήτησης ελπίδα μας είναι αυτό που ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν ξεκινήσει να συνεχιστεί και να μπορέσουν να ε, καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη νέα πρόταση οδηγίας την οποία θα μελετήσουμε με μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ. Σας συγχαίρω για τον διορισμό σας ως Αντιπροέδρου της Οργανισμού για τον Δικαιώμα των Παιδιών. Κύριε Μωράης, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το επίτευγμα της κυρίας Χέτ και της κυρίας Μπάουερ σήμερα ήταν, παρόλο που μιλάμε πολύ αργά, ήταν ότι ήρθαν εδώ απόψε και συνάντησαν τον κύριο Μπαρό και τον νέο, τον νέο εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας και να τους ακούσουν να χρησιμοποιούν όρους όπως αποφασιστικότητα, φιλοδοξία, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άξιζε να είμαστε εδώ τόσο αργά για να τα ακούσουμε αυτά. Διότι υπήρξαν πολλοί σήμερα στην αίθουσα συμπεριλαμβανομένων και των συντακτριών που αντιλαμβάνονται πόσο περίπλοκο είναι το σύγχρονο αυτό φαινόμενο και αντιλαμβάνονται επίση ότι αναμένεται από του πολίτε, οι πολίτε περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει αυτή τη σύγχρονη μάστιγα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σύντομα την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριο Βαροκυρία Μάλστρομ, ανταποκρίθηκε θετικά στι προτάσει μα για τον, συντονιστεί στον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται βήματα προς τα μπρος η κλίμακα του φαινομένου, όπως είπε η Άννα Χέντ, σημαίνει ότι πρέπει να ενεργήσουμε με αποτελεσματικότητα. Εφόσον πρόκειται για τόσο περίπλοκο φαινόμενο που αγγίζει τόσους πολλούς τομείς, οργανωμένο έγκλημα, υποχρεωτική καταναγκαστική εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, γυναικών κλπ. Ο κύριος Μπαρό αναφέρθηκε σε πάρα πολλά πράγματα που θα θέλαμε να γίνουν πραγματικότητα αν αποτελέσουν ένα πακέτο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταλήξουμε σε μια αποφασιστική πολιτική η οποία για τους πολίτες θα είναι ένα σχέδιο δράσης. Οι πολίτες γνωρίζουν τη μάστιγα της εμπορίας ανθρώπων αλλά δεν βλέπουν καμία συγκεκριμένη πρόταση, καμία συγκεκριμένη προσπάθεια. Με τα χαράς άκουσα την ε, υποψήφια επίτροπο ε, την κυρία Μάλστρομ να μας λέει ότι σύντομα θα υπάρξουν αυτά αποτελέσματα και την Ισπανική Προεδρία που μας είπε ότι θα ληφθούν δραστικά μέτρα. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν για να αποδείξουν την ε, αποφασιστικότητα όλων μας για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Παρόλο που είναι αργά πρέπει πλέον να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη και σε αυτό μας βοήθησαν οι συντάκτριε με την ερώτησή του, Η κυρία Χίρ, επόμενη ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους που υπέβαλαν αυτή την ερώτηση. Πρόκειται για μια σοβαρή δέσμευση, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, πρόκειται, αν θέλετε, για ένα το αδίκημα. Τα στοιχεία που διαθέτουμε από τη Europol μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει βελτίωση, υποχώρηση του φαινομένου. Αντίθετα αυτή η καταναγκαστική εργασία και η εκμετάλλευση δυστυχώς αυξάνεται. Χρειάζεται λοιπόν άμεση δράση, είναι επίγον το θέμα και πιστεύω ότι αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς και αποτελεσματικοί στη δράση μας θα πρέπει να έχουμε μια συλλογική και ενσωματωμένη δράση σε όλους αυτούς τους τομείς της εκμετάλλευσης. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι η συνειδητοποίηση στην Ευρώπη του τι συμβαίνει, ότι αυτή η εμπορία ανθρώπων λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης και σε όλα τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει επίσης να πούμε ότι όπως κάναμε και στη Γερμανία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, με μηνύματα και συγκεκριμένες δράσεις τι ακριβώς συμβαίνει, να συνειδητοποιήσει το κοινό και να ευαισθητοποιηθεί. Ένα δεύτερο σημείο, η προστασία των θυμάτων. Πιστεύω τα άτομα αυτά που ζουν αυτές τις δραματικές συνθήκες θα πρέπει να τους προσφέρουμε μία ψυχολογική, ή ιατρική υποστήριξη έτσι ώστε να μπορέσουν όσο ζουν στις χώρες μας να ξεκινήσουν ε, μια νέα ζωή είτε στη νέα τους χώρα είτε να μπορέσουν να γυρίσουν στις χώρες τους. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα σε μια Ολλανδική εφημερίδα κυκλοφόρησε ένα άρθρο για έναν καλλιεργητή σπαραγγιών, μια ε, καλλιεργήτρια ε, σπαραγγιών, διότι θεωρήθηκε ότι ήταν υπεύθυνη δουλεμπορίου κατά Ρουμάνων υπηκών. Βλέπουμε ότι το θέμα αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ολοκληρωμένη πολιτική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων δεν μπορεί να περιορίζεται στη σύλληψη κάποιου δουλεμπόρου δεν μπορούμε να ε, διώκουμε τους δράστες αλλά πρέπει να δείξουμε ενδιαφέρον και για τα θύματα αυτών των εγκληματικών ενεργειών. Τα θύματα δεν πρέπει ποτέ να έχουν την εντύπωση ότι είναι μόνα τους εγκαταλειμμένα. Δεν τους έχουμε εγκαταλείψει, δεν τους εγκαταλείπουμε. Τους, πρέπει να τους παρέχουμε όλη την κοινωνική, ιατρική, οικονομική, δικαστική, νομική βοήθεια και να τους καταβάλουμε και αποζημιώσεις ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθεί αυτό στη νέα οδηγία. Ο κύριος Μπαρό και ο κύριος Λόπες Γκαρίγκο είπαν πολύ σημαντικά πράγματα. Ο Επίτροπος συγκεκριμένα είπε ότι εκείνοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ε, ατόμων που είναι θύματα δουλείας πρέπει να καταδικάζονται επίσης. Αυτό θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο. Διερωτώμε ωστόσο πώς θα, βοηθήσουμε, πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα θύματα εάν ε, ποινικοποιούμε την εργασία τους. Πώς θα βοηθήσουμε τα άτομα αυτά αν ανησυχούν ότι θα διωχθούν ποινικά λόγω της εργασίας που έχουν αναλάβει. Η εμπορία οι πράσινοι πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων μια μόνιμη άδεια παραμονής, κάτω από ορισμένε προϋποθέσεις βεβαίως, για να ξέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να διωχθούν πίσω στη χώρα από την οποία ξεκίνησαν όλα. Ξέρουν επίσης ότι μπορούν να καταγγείλουν και να υποβάλουν μήνυση ε, κατά των δουλεμπόρων υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, χωρίς κανένα κίνδυνο να σταλούν πίσω στη χώρα όπου έπεσαν θύματα των δουλεμπόρων. Ελπίζω λοιπόν ότι η νέα ε, οδηγία πλαίσιο θα εξασφαλίσει περισσότερα δικαιώματα στα θύματα και θα σου εγγυηθεί ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό ελπίζω να δω στο κείμενο που θα μας παρουσιάσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Τσιόμπρο για ένα λεπτό. Κύριε Τσόπρο, ευχαριστώ πολύ. Είναι πονίδιστο το γεγονός ότι η σύγχρονη Ευρώπη που απολαμβάνει την ελευθερία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει γίνει ένας χώρος δουλείας για τόσους πολλούς ανθρώπους και ένας χώρος κατάχρησης και εκμετάλλευσης. Είναι θλιβερό διότι πολλές φορές αφορά ευάλωτα άτομα, δηλαδή γυναίκες και παιδιά. το δικαστικό σύστημα και εγώ ως εισαγγελέα στην ε, Πολωνία ε, υπήρξα μάρτυρας πολλών τέτοιων δικαστικών διαδικασιών και ε, πραγματικά διαπιστώνω ότι τα εγκλήματα δεν έχουν φραγμούς. Το ίδιο ισχύει και για την εκμετάλλευση των παιδιών και τη σύγχρονης δουλείας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει αρχές στα κράτη-μέλη να είναι κεντρικές και επαγγελματικές και να ενισχύεται η συνεργασία. Θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ σημαντικός ρόλος και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γνωρίζουμε ότι η εμπορία ανθρώπων είναι η ευθύνη ε, οργανώσεων ε, και θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ποινές για αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσουμε να κατασχέσουμε τα εισοδήματα των ανθρώπων που ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων. Η κυρία Έρνστη, 1,5 λεπτό. Η εμπορία ανθρώπων είναι πραγματικά σημερινός τρόπος δουλείας. Η χειρότερη μορφή αυτής της δουλείας είναι με θύματα ανήλικα παιδιά. Και πραγματικά η πολιτική μου ομάδα θεωρεί ότι πρέπει η Επιτροπή να αντιδράσει άμεσα και με επίγοντα τρόπο. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο την, ε, το εμπόριο ανθρώπων, θα πρέπει πραγματικά να αντιδράσουμε ξεκινώντας από την πρόληψη. Δεν είναι δυνατόν αυτό το φαινόμενο να καταπολεμηθεί μόνο με κυρώσεις και ποινές. Χρειάζονται πολύ συγκεκριμένοι κανονισμοί και ρυθμίσεις όσον αφορά βεβαίως και τις κυρώσεις του φαινομένου αυτού. Χρειάζεται προστασία, προστασία των θυμάτων μετά από μια συγκεκριμένη ποινική διαδικασία η οποία θα έχει εναρμονιστεί. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τις απειλές και τις κατηγορίες. Είναι απαραίτητο σήμερα η προστασία να ξεκινήσει με μακροχρόνιους στόχους. Και η προστασία των θυμάτων δεν θα πρέπει μόνο να ε, στοχεύει τα παιδιά. Τα παιδιά βεβαίως είναι τα πιο ευάλωτα θύματα αυτής της εκμετάλλευσης. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν δεσμευτικές πολιτικές όσον αφορά την προστασία, την πρόληψη και να συμπεριλαμβάνονται και αστυνομικοί και δικαστές και ψυχολόγοι. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα ε, μέτρα που προτείνατε. Ο κύριος Μποργέτσιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα σήμερα κατά τη διάρκεια της ακρόασης της υποψήφιας επιτρόπου μια πολύ συγκεκριμένη δέσμευση για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων και εδώ σήμερα με χαρά ακούω μια ομόφωνη άποψη. Δεν υπήρχε ομόφωνη άποψη όταν ε, πολλά χρόνια πριν κάποιοι εδώ στα έδρανα, μεταξύ των οποίων και εγώ, ε, κατάγγελαν τους ε, κινδύνους που θα προέκυπτε από τη μαζική μετανάστευση και τα δίκτυα τα εγκληματικά τα οποία εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και τον κίνδυνο εκμετάλλευσης ανθρώπων αλλά και των οργάνων τους. πλέον σήμερα όλοι αναγνωρίζουν αυτό το φαινόμενο και θα πρέπει να χαιρόμαστε για το γεγονό γεγονός ότι είναι πλέον ομόφωνη η φωνή και να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το αίτιο είναι πάντα ε, το ίδιο. Το αίτιο έχει πάντα ένα όνομα η διεύρυνση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι εγκληματικές οργανώσεις, οι τοπικές, οι, ευρωπαϊκές, οι ευρωπαϊκές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι πλέον έχουμε και ε, δίκτυα τα οποία διαχειρίζονται και έξω ευρωπαϊκά ε, σε εγκληματικές οργανώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από εκεί, να λάβουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι αυτό το τόσο φοβερό, σοβαρό και επονίδιστο ε, φαινόμενο είναι συνέπεια της παράνομης μετανάστευσης η οποία γίνεται μαζικά και δεν ελέγχεται καταλήλως. Η Ευρώπη πρέπει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Η κυρία Ντότς, απουσιάζει ο κύριος Παπα-Νικολάου. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τις συντάκτηρες της πολύ σημαντικής αυτής ερώτησης ζούμε σε ένα σύγχρονο κόσμο που θα περίμενε κανείς ότι τα φαινόμενα εμπορίας ανθρώπων θα είχαν εκλείψει από την κοινωνία μας. δυστυχώς όμως τα νούμερα μας διαψεύδουν και επιτρέψτε μου να παραθέσω μερικά. περισσότερο από ένα εκατομμύριο 800.000 παιδιά και νέοι άνθρωποι εκτιμάται ότι πέφτουν κάθε χρόνο θύματα του τράφικινγκ παγκοσμίω. 270.000 θύματα ε, περιγράφουν τα ηνωμένα έθνη ότι έχουμε στην ευρωπαϊκή ένωση. μόνο στην ελλάδα οι εκτιμήσει ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων εμπορίας με σκοπό την πορνεία σε 40.000 ετησίω συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών χωρίς όμως να περιλαμβάνουμε τις άλλες μορφές τράφικινγκ. οι δύο αδυναμίες οι πιο βασικέ που θα ήθελα να επισημάνω χωρί να υποτιμώ τι άλλε παραμέτρου είναι οι εξή πρώτον το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτού του εγκλήματο που είναι διασυνοριακό και επιτείνεται από τη λαθρομετανάστευση όπω σωστά υπόθηκε δεν είναι επαρκέ και γι' αυτό είναι ανάγκη να επιταχύνουμε το βήμα μα προ μια ολιστική προσέγγιση και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η οδηγία που αναμένουμε όπω πολύ σωστά ανεφέρθη. δεύτερον ιδιαίτερο κενό εντοπίζεται στην προστασία των θυμάτων και ιδίως στο ζήτημα των υποστηρικτικών δομών. είναι λοιπόν απαραίτητο και χαίρομαι πολύ που το άκουσα αυτό από την ισπανική προεδρία να διατεθούν πόροι και υποδομές προκειμένου να βελτιωθούν οι όποιες υπάρχουσες υποδομές και να δημιουργηθούν και νέες και βεβαίως να εκπαιδευτεί και κατάλληλα ε, το προσωπικό που μπορεί να προσφέρει μια τέτοια υποστήριξη η σύγχρονη αυτή μορφή δουλεμπορίου δεν πρέπει και δεν μπορεί να έχει καμία θέση σε μια ευρωπαϊκή ένωση που ως βασική της συνιστόσα έχει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Κώστα, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι εμείς σήμερα ασχολούμαστε με ένα θέμα όπως αυτό, με την πολύ σημαντική προφορική ερώτηση, για την οποία θέλω να ευχαριστήσω τις συντάκτριες, ε, αλλά και την ε, πολύ καλή συνεργασία που υπήρχε από όλες τις πολιτικές ομάδες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα πολύ σοβαρή δέσμευση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Προεδρία του Συμβουλίου και εύχομαι πραγματικά αυτή η νέα οδηγία να ξεκινήσει ε, υπό το φως των ε, ε, κατευθυντηρίων γραμμών που νομίζω ότι συμμερίζονται όλοι στο θέμα αυτό. Ξέρετε ότι είναι πολύ περίπλοκα τα θέματα τα οποία πρέπει να αναλύσουμε. Μιλάμε περίπου για 300.000 ε, άτομα, ε, περίπου το 90% είναι γυναίκες και παιδιά ε, που είναι θύματα εμπορίες και δυστυχώς υπήρξε αύξηση τα τελευταία χρόνια. Και θα πρέπει λοιπόν να γίνει και ένα σημαντικό βήμα βάσει και των νέων αρμοδιοτήτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει και των όσων εγκρίμενα με ήδη στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης για να έχουμε κάποιες καινοτομίες Έγινε ένα τεράστιο άλμα όταν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκε ο κανόνας που ισχύει στην Ιταλία ήδη από το 1998, το δικαίωμα παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά θα πρέπει να σταθούμε κυρίως στα θέματα για θέματα προστασίας, κοινωνικής ενσωμάτωσης, ε, θέσεων εργασίας, προστασία ε, και τιμωρία για τον πελάτη ε, και επίσης ε, ποινές ε, και κυρώσεις όπως είπατε και εσείς κύριε Επίτροπε οι οποίες θα πρέπει να εναρμονιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης ζητάμε να αξιολογηθεί η συνένεση των θυμάτων σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης, διότι τις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει εκβιασμός και να υπάρχει και συγκεκριμένη μέρημνα όχι μόνο για τους ανηλίκους, αλλά να υπάρχουν και μορφές υποστήριξης για άτομα τα οποία φτάνουν στην Ευρώπη, που έχουν ήδη υποστεί εμπορία ε, καθ' τη διαδρομή, την τραγική διαδρομή την οποία διανύουν προκειμένου να φτάσουν στις ακτές μας και στα εδάφη μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παρβανόβα λεπτό. Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ του συγγήτριες, την Ισπανική Προεδρία, την Επιτροπή για τη δέσμευση να βρουν μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Όταν μιλάμε για εμπορία ανθρώπων είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη την ε, δημιουργία ε, μιας πλατφόρμας ενός βήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της δράσης των κρατών μελών για την προστασία των θυμάτων αυτής της εμπορίας, αυτού του σύγχρονου δουλεμπορίου. Θα πρέπει επίσης να καθιερωθεί και ένας συντονιστής, ένας συντονιστής μια συντονιστική υπηρεσία ώστε όλα τα κράτη-μέλη να ακολουθούν αντίστοιχη προσέγγιση για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος να ληφθούν προληπτικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τη στενή συνεργασία μεταξύ ε, των κρατών μελών και την προσώπων της κοινωνίας των πολιτών, να οργανώσουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και να δώσουμε όλη την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη στα θύματα αυτής της εμπορίας. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμός και στρατηγικές δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθηθούν τα επιμέρους κρατημέλη να καταπολεμήσουν αυτή τη σύγχρονη μάστιγα. Ο κύριος Γιανακουδάκης για ένα λεπτό. Κυρία, συγγνώμη. helpless victim of some dominating ένα απελπισμένο θύμα αυτής της ε, κυριαρχίας. Ε, αυτή δεν είναι μορφή δουλείας, είναι, ε, δεν είναι μορφή εμπορία, συγγνώμη, είναι μορφή δουλείας. Η εμπορία ανθρώπων είναι δουλεία και εκμετάλλευση ανθρώπων, ανδρών, γυναικών και παιδιών είναι αδίκημα η απόλυτη ένδια, η διάλυση της οικογένειας, η εσωτερική οικογενειακή βία συνεισφέρουν ορισμένες φορές στην εμπορία ανθρώπων. Στην Ευρώπη ε, εκτιμούμε ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα και με, ε, και η πλειονότητά τους είναι ε, παιδιά. Οι υπηρεσίες εφαρμογή της νομοθεσίας, οι συνοριοφύλακες, οι αστυνομικές δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν. Ε, πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί για την υποστήριξη. Ε, οι θεσμοί θα πρέπει να είναι πολύ ισχυροί, να κατευθύνονται από τα κράτη-μέλη και να υποστηρίζονται από τα κράτη-μέλη. Η κυρία Σβένσον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν χτυπήσουμε τη ζήτηση θα πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει ζήτηση για παιδιά, για σεξουαλικές υπηρεσίες, τότε δεν θα εξαφανιστεί και η εμπορία ανθρώπων. Η ζήτηση είναι η λέξη κλειδί λοιπόν όταν μιλάμε για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο ζουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες φτώχειας και ως εκ τούτου είναι πολύ εύκολα, πέφτουν πολύ εύκολα θύματα εκείνων που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να περιορίσουμε, όπως είπα, τη ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες και να εφαρμόσουμε και μέτρα πρόληψης βελτιώνοντας παραδείγματος χάρη τις συνθήκες διαβίωσης ε, στις περιοχές του κόσμου από όπου γίνεται συνήθως η, επιλογή των θυμάτων. Εγώ και η ομάδα μου ευχαριστούμε την κυρία Χέτ και την κυρία Μπάουερ και τους συναδέλφους της Αρμόδιας Επιτροπής. Ωστόσο θα ήθελα ε, να δω κάποιες διαφοροποιημένες προτάσεις για το πώς μπορούν να υποστηριχθούν τα θύματα και να τους παρασχεθεί βοήθεια. Χρειαζόμαστε ένα ευρύ φάσμα μέτρων που θα ποικίλουν ανάλογα για το αν πρόκειται για σεξουαλική εκμετάλλευση ή καταναγκαστική εργασία. Χρειαζόμαστε διαφορετικά μέτρα και ε, πολιτικές για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων. Χιμένες για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα με μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε περίπου 270.000 άτομα τα οποία υπήρξαν θύματα ε, εμπορίας ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τέτοια στοιχεία είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί κυρίως στην προστασία των θυμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή ε, στην κατάσταση των ε, γυναικών και των παιδιών που είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες. Δεν μπορούμε να διαφορούμε σε αυτό, μπροστά σε αυτή την παράσταση σεξουαλικής εκμετάλλευσης η οποία εκτιλήσεται μπροστά στα μάτια μας. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ την υποστήριξη του Κοινοβούλιο διότι η συνδρομή προς τα θύματα θα πρέπει να γίνεται άνω και θα πρέπει να ε, είναι και οι ποινές πολύ πιο σοβαρές όπως είπε και ο κύριος Μπαρό. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ισπανική Προεδρία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν όλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που έχουν στη διάθεσή τους τόσο την κείμενη όσο και τη μελλοντική για να προστατεύσουν τα θύματα της ε, εμπορίας θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα προστασίας των θυμάτων. Το είχα ζητήσει και από την Ισπανική Προεδρία κατά τη συζήτηση για το πρόγραμμα της Στοχόλμης και ε, το θέμα της ε, οδηγίας θεωρώ ότι θα είναι αποτελεσματικό για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Ε, η Ισπανική Προεδρία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου αυτό το ένταλμα να έχει αποτελεσματικά ε, μέτρα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να μπορέσουμε να δράσουμε έτσι μπροστά σε κάποια από τα πιο σοβαρά προβλήματα ε, της κοινωνίας μας με πολύ συγκεκριμένε λύσεις όπως είναι το θέμα της εμπορίας ανθρώπους. Να μην μένουμε μόνο στα λόγια αλλά ε, να κάνουμε και πράξεις. Το οφείλουμε στα θύματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπένοβα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στις εισηγήτριες Head και Bauer οι οποίες με κάλυψαν πλήρως αυτό το θέμα και θα ήθελα τώρα να προσθέσω μερικές προσωπικές σκέψεις. Δεν γνωρίζουμε πάντοτε ποια είναι η έκταση αυτού του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων. Είναι ίσως ο πιο κερδο, η πιο κερδοφόρα παράνομη δραστηριότητα στον κόσμο που πλήττει κυρίως γυναίκες και παιδιά. Η απάντησή μας λοιπόν πρέπει να είναι μαζική, η καταπολέμηση αποτελεσματική και να εστιαστεί σε όλη την έκταση του, σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Το σύγχρονο, η σύγχρονη αυτή μορφή δουλείας υπάρχει σε περιοχές όπου υπάρχει ανεργία, ε, πολιτική αστάθεια, φτώχεια κλπ. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προσφέρουμε μια αξιοπρεπή ζωή σε αυτά τα άτομα για να μην είναι πλέον θύματα αυτής της παράνομης δραστηριότητας και πρέπει να προβλεφθούν και πιο αυστηρές κυρώσεις κατά των σύγχρονων αυτών δουλεμπόρων. Οι χρήστε των υπηρεσιών πρέπει και εκείνοι να τιμωρούνται με παραδειγματικές ποινές κυρίως κατά των δουλεμπόρων. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε στενή συνεργασία με την Eurojust, την Europol και την Frontex. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο θέμα της σύγχρονης δουλείας αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι η πώληση σαν ένα κομμάτι κρέας ανθρώπινων όντων, ανδρών, γυναικών και ανήλικων παιδιών. Πρόκειται για άτομα των οποίων παραβιάζονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τα οποία γίνονται θύματα εκμετάλλευσης. Φυσικά, και αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να καταπολεμήσουμε την ίδια ώρα και την προσφορά και την ζήτηση. Στη χώρα μου ο νόμος απαγορεύει την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών και η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι και 10 χρόνια φυλάκισης. Είναι πολύ σημαντικό να ενσωματωθεί στο κείμενο αυτό και το θέμα της απαγόρευσης της πώληση των ανθρώπινων όντων και της εμπορίας τους. Πριν από 150 χρόνια καταργήθηκε η δουλεία στην Αμερική. Βλέπουμε όμως ότι τα φαινόμενα αυτά συνεχίζουν. Γι' αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Επίτροπε, Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά, οι εκπρόσωποι Πρασίνων πολύ σωστά είπαν ότι αυτό το θέμα, η εμπορία ανθρώπων, δεν είναι εξωτερικό πρόβλημα το οποίο εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εσωτερικό πρόβλημα της Ένωσης. Οι πολίτες της χώρας μου πολλούνται, έχουν πολιθεί σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα και κατά την άποψή μου πρέπει να ενεργήσουμε με αλληλέγγυο και ενωμένο τρόπο, όχι μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών. Και θα, θα ήθελα να σας θυμίσω γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από αρκετά χρόνια, όταν η Ιταλική αστυνομία και η Ιταλική διοίκηση αντέδρασε σε κάποια μηνύματα από την Πολωνία Μιλάμε για περιπτώσεις εμπορίες ανθρώπων. Ε, μιλάμε για Πολωνούς εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν θύματα εκμετάλλευσης. Η κυρία Ρόιταβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε χρόνια πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι είναι θύμα εκμετάλλευσης ε, σεξουαλικής εμπορίας. Μόνο 1.005 περιπτώσεις έχουν καταλήξει στο δικαστήριο παρά το γεγονός ότι είχαμε τεράστιο αριθμό θυμάτων. Αυτό καταδεικνύει ότι τα έσοδα από την εμπορία ανθρώπων είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα για, από τα ναρκωτικά. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση επεκτείνεται προς Ανατολάς, αυτό το οργανωμένο έγκλημα αυξάνεται. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια συντονισμένη στρατηγική και να ληφθούν συγκεκριμένα βήματα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να είναι ενάντια στην εναρμόνιση της νομοθεσίας. Ε, στρέφομαι προς την Ισπανική Προεδρία και του ζητώ να οριστικοποιήσουν τις ομιλίες μεταξύ κρατών ομιλών για τον καθορισμό των συγκεκριμένων ποινών και κυρώσεων και η νέα οδηγία την οποία περιμένουμε θα πρέπει να είναι πιο αποδοτική και θα πρέπει να μειώσει τη ζήτηση για παράνομη, ε, σε, παράνομες σεξουαλικές υπηρεσίες. Το θέμα της εκμετάλλευσης ε, των παιδιών είναι σε αύξηση. Είμαστε πάνω από το 20% ε, για τα παιδιά και θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση και για τα παιδιά και για τους γονείς τους. Ξέρετε ότι μόνο το 4% των παιδιών ε, που υπήρξαν θύματα εκμετάλλευσης έχουν παραδεχθεί ότι χρησιμοποιήθηκε το διαδικτύο για να ε, κανονιστεί μια συνάντηση με το παιδί τους. Κατά τη διάρκεια του 2009 υπήρχαν πάμπολες ε, ιστοσελίδες που ανακαλύφθηκαν στο διαδίκτυο, οι οποίες προήγαγαν τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μειώσουμε τη ζήτηση και να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το θέμα της εμπορίας ανθρώπων. Ζητώ λοιπόν να παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κατάλληλο πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Η κυρία Γκόγκς δεν είναι εδώ. Η κυρία Τόμσεν, λοιπόν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη συζητήτρια για αυτή την πολύ σημαντική πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα ένα τεράστιο θέμα, μια μεγάλη πρόκληση που είναι η καταπολέμηση των ανθρώπων, η καταπολέμηση του εμπορίου των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι σήμερα οι κυρώσεις είναι πάρα πολύ ελαστικές και καθόλου αυστηρές σε σχέση με άλλου είδους παρόμοια φαινόμενα και εγκληματικές δραστηριότητες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι τα θύματα αυτής της εκμετάλλευσης δεν μπορούν να εγκαταληφθούν σε αυτούς που τους εκμεταλλεύονται και θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα προστασίας και την ίδια ώρα θα πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα η σεξουαλική προσφορά υπηρεσιών και η καταναγκαστική εργασία. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που η Επιτροπή ασχολείται αυτή τη στιγμή με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα πρόσφατα γεγονότα στη Λιθουανία που μια οργάνωση εμπορία ανθρώπων συνελήφθη έδειξαν και πάλι ότι αυτές οι μορφές εγκλήματος είναι ένα ευρύτατα διαδεδομένο φαινόμενο που εντείνεται και διονγκώνεται σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης. Τα περισσότερα θύματα είναι δυστυχώς γυναίκες και παιδιά που λόγω φτώχειας η εμπορία ανθρώπων είναι ένα φρικτό έγκλημα μια, μια ταπείνωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με τις τρίτες χώρες προκειμένου να, και να εξασφαλιστεί ένας μόνιμος διάλογος με τις ΜΚΟ και να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει έναν συντονιστή για τα θέματα εμπορίας ανθρώπων. Στα θύματα που να δοθεί όλη η αναγκαία προστασία και βοήθεια και η δυνατότητα ενσωμάτωσης στις ε, κοινωνίες των χωρών υποδοχής. Αυστηρές κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν κατά των ε, ε, υπεύθυνων αυτών των εγκλημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια αυτής της προφορικής ερώτησης και θα ήθελα να πω και εγώ ότι το εμπόριο ανθρώπων είναι μια πάρα πολύ κερδοφόρα δραστηριότητα. Οι στατιστικές μας δείχνουν ότι 700.000 ή 1 εκατομμύριο θύματα υπάρχουν στον τομέα αυτό και ένας μεγάλος αριθμός αυτών βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε και εμείς από την Επιτροπή να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο με πολύ αυστηρότερα μέτρα να τιμωρούνται όχι μόνο οι εκμεταλλευτές και οι διοργανωτές αυτών των δραστηριοτήτων, αλλά και οι χρήστες. Επίσης, την ίδια ώρα θα πρέπει να υπάρξουν και συνοδευτικά μέτρα προστασίας των θυμάτων και τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να προσέξουν για να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κυρώσεων και της αντιμετώπισης αυτών των ποινικών πράξεων. Τα θύματα θα πρέπει επίσης ιδιαίτερα να προστατευτούν, ιδιαίτερα όταν είναι ανήλικα παιδιά. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα απαγορευθούν αυτές οι δραστηριότητες από τις χώρες μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της εμπορίας των ανθρώπων να συζητηθεί Δυστυχώς, στην σημερινή κοινωνία των δυτικών χωρών, κυρίως γυναίκες είναι θύματα αυτού του εμπορίου. Σκέφτομαι και την πορνεία, αλλά και τα θύματα που είναι παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε τη δράση μας προς αυτές τις ευάλωτες κατηγορίες πολιτών και αυτό βεβαίως ε, μου υπενθυμίζει ότι θα χρειαστούν και επιπλέον μέσα πόροι. Δεν μπορούμε βεβαίως να κάνουμε τίποτα αν δεν ε, γίνουν αυστηρότερες οι ποινές, αν δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας και γι' αυτό χρειάζονται πόροι έτσι ώστε να μπορέσουν τα άτομα αυτά να επανενσωματωθούν στην κοινωνία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανήλικα θύματα και να μπορέσουν με ένα νόμιμο τρόπο να ενσωματωθούν στην αγορά των χωρών μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή δράση επί του θέματος έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και γι' αυτό χάρηκα που άκουσα τις παρατηρήσεις του κυρίου Γκαρίντο για το θέμα αυτό και για τα παιδιά. Η υποψήφια επίτροπος μας είπε η κυρία Μάλστρομ σήμερα το πρωί ότι σκοπεύει να παρουσιάσει μια οδηγία ω προτεραιότητα επί του θέματος. Θα ήθελα να δείτε και τα συστήματα υποστήριξης για τα θύματα, κυρίως τις ανάγκες ε, των παιδιών που είναι θύματα εμπορία, που είναι πολύ διαφορετικές από τους ενήλικες που είναι θύματα εμπορία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρσι 325 παιδιά ήταν ε, ύποπτα ως θύματα εμπορίας και Πρόκειτο για ε, πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ε, υπήρξαν θύματα εμπορίας εντός του, της επικράτειας. Υπάρχουν παιδιά στην ίδια μου την περιοχή που υπήρξαν θύματα εμπορίας, αλλά ε, διαπιστώσαμε ότι ακόμα και αν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα των Κοινωνικών Υπηρεσιών, πολλά παιδιά εξαφανίζονται γιατί είναι ακόμα υπό τον έλεγχο των ανθρώπων που τα εκμεταλλεύονται και θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να τα ξαναεμπορευθούν. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άτομα τα οποία είναι θύματα εμπορία είναι χωρί φωνή, είναι ευάλωτα και χρειάζεται να μιλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξ ονόματό του και να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να τα φροντίσει κάποιο. ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τα αδικήματα κατά γυναικών και παιδιών. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο όπως μας δείχνουν οι αριθμοί και τα στοιχεία διαρκώς αυξάνεται και παίρνει νέες διαστάσεις. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των εκμεταλλευτών λειτουργεί από τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης ότι τα θύματα βεβαίως δεν είναι απλώς θύματα που έρχονται από τρίτες χώρες αλλά από και τις ίδιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν βεβαίως να ελέγξουμε τα εξωτερικά μας σύνορα για να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό, κάτι το οποίο σήμερα δεν γίνεται. Επίσης βλέπετε ότι πρόκειται για έναν τουρισμό εγκληματικό με λεωφορεία συνήθως μετακινούνται τα θύματα αυτής της εκμετάλλευσης και από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία της Europol και της Frontex οι συνοριακές αυτές περιοχές δεν ελέγχονται, τα σύνορά τους είναι ανεξέλεγκτα, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια νέα αντιμετώπιση. Θα ήθελα πράγματι να σας ευχαριστήσω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η προφορική ερώτηση μας δείχνει ότι ο κίνδυνος να γίνει κανείς θύμα αυτής της εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες και τα παιδιά. Βλέπουμε από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε ιδιαίτερα τα παιδιά και τα ανήλικα θύματα, ενημερώνοντας και προλαμβάνοντας αυτήν την εγκληματική δράση. Επίσης, όταν ένα παιδί είναι θύμα αυτής τη εκμετάλλευση. θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσει να προστατευθεί, να βοηθηθεί και να ξαναενσωματωθεί στην κοινωνία. Η πρόληψη όμως είναι πολύ σημαντική. Η πρόληψη θα πρέπει να λάβει χώρα στις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτά τα παιδιά, αυτά τα ανήλικα θύματα και προς τους γονείς και τις οικογένειές. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να εξετάσουμε τρία θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία και χρειάζονται προσοχή. Δεν υπάρχουν αρκετοί εγκληματίε που προσάγονται στη δικαιοσύνη παρόλο που το φαινόμενο της εμπορίας ε, ανθρώπων αυξάνεται διαρκώς. Το δεύτερο θέμα είναι τα θύματα δεν ε, την χάνουν της δέουσας βοήθειας και αποζημίωσης. Λόγω της έκτασης αυτού του φαινομένου στην Ευρώπη, ελάχιστα κράτη-μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα. Τρίτον, η κατάσταση δεν παρακολουθείται και ελέγχεται ε, αποτελεσματικά. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες ώστε να ε, ε, καταπολεμηθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο η εμπορία ανθρώπων. Τελείωσε η διαδικασία του Catch the Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Λόπτης Γκαρίντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση κατέδειξε ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός πολύ σοβαρού προβλήματος, ένα πρόβλημα το οποίο αποτελεί τεράστια πρόκληση και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα διότι έγινε αυτή η συζήτηση την ημέρα της πρώτης μου παρέμβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι τιμή αδιαμφισβήτητα για μένα και ε, βρέθηκα εδώ σε αυτές τις δύο πολύ σημαντικές συζητήσεις που έγιναν απόψε για ε, εδώ σε αυτό το πολύ σημαντικό και ισχυρό κοινοβούλιο. Το τεράστιο αυτό πρόβλημα δεν μπορούμε απλώς να το αναφέρουμε ή απλώς να το σκεφτόμαστε, θα πρέπει να πολεμήσουμε με σθένος, διότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόβλημα και οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολύ ισχυρέ. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται τεράστια πολιτική βούληση για το θέμα αυτό. Σήμερα αποδείχθηκε ότι υπάρχει τεράστια πολιτική βούληση και εγώ θα σας πω ότι η Ισπανική Προεδρία θα την αποδείξει και αυτή την ε, ε, πολιτική βούληση για να μπορέσει να συνεργαστεί και να ε, προσπαθήσει να εξεύρει μια λύση επί του θέματος μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από την Ευρώπη αυτό το πρόβλημα. Ε, ακούσαμε ότι το φαινόμενο υπάρχει και στην Ευρώπη. Ε, οι κύριοι Παπα-Νικολάου, η κυρία Παρβανόβα κατέδειξαν το διαμεθοριακό χαρακτήρα αυτού του θέματος υπάρχει στην Ευρώπη και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από την Ευρώπη. Επαναλήφθηκε πολλές φορές, θα το επαναλάβω και εγώ άλλη μία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας παρουσιάσει μία οδηγία για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε υπό αυτό το πρίσμα. Νομίζω ότι πολύ σωστά το είπε και η κυρία Ρόιτοβα στην παρέμβασή της. Και θεωρούμε ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες που θα πρέπει να ε, ε, επισημάνουμε είναι ε, η εργασία που θα πρέπει να γίνεται από πλευρά Ευρώπη για την προστασία των θυμάτων πρώτον. Η προστασία των θυμάτων είναι το πιο βασικό ζήτημα και είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε τι περισσότερε φορέ σήμερα. Ε, οι συντάκτηρε της ε, προφορική ερώτηση, η κυρία Αντζελίλη και πολλοί άλλοι από τους προλαλήσαντες επεσήμαναν πόσο σημαντικό είναι το θέμα τη προστασία των θυμάτων που τείνουν να είναι γυναίκε και παιδιά, οι πιο ευάλωτε ομάδες, το ανέφεραν ε, και άλλες κυρίες απόψε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την προστασία των θυμάτων. Ένα ένταλμα προστασίας των θυμάτων που αποτελεί προτεραιότητα για την Ισπανική Προεδρία. Πρώτον λοιπόν προστασία των θυμάτων. Δεύτερον, μια πάρα πολύ αυστηρή τιμωρία για τους εμπόρους. Πολύ σωστά το είπε κάποιος από τους ομιλητές. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε, επαναλαμβάνω, το θέμα της ζήτησης αυτών των υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει μεν να εργαστούμε πολύ σκληρά για να το κάνουμε, αλλά δεν πάβει να είναι με ένας πολύ σημαντικός άξονας του προβλήματος. Έτσι έχουμε τις τρεις βασικές διαστάσεις ε, και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση ε, για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, για το οποίο επαναλαμβάνω κύριοι και κυρίες Ευρωβουλευτές, η, η Ισπανική Προεδρία είναι και θα είναι συνεχώς δεσμευμένη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Τελευταίο ο ο κύριο Μπαρό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση πράγματι έριξε φω για την προεκτιμασία της μελλοντικής οδηγίας την οποία σκοπεύει να παρουσιάσει κατά την Άνοιξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε ο Κλοντ Μωράς, θα πω και εγώ ότι πρέπει να αγωνιστούμε με τα μέσα τα πιο σύγχρονα που διαθέτουμε κατά αυτής της μάστιγας. που και αυτή χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα μέσα για να εξαλείψουμε κάθε μορφή εκμετάλλευσης. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν τρεις πυλώνες ε, η, τα θύματα, η βαρύτητα των κυρώσεων και το θέμα της ζήτησης. Θα επιμείνω στην προστασία των θυμάτων, διότι στην απόφαση πλαίσιο είχαμε ήδη συζητήσει την προστασία σε όλα τα θύματα ανεφόρων, την δικαίωμα σε νομική ε, βοήθεια και στη μελλοντική οδηγία θα ασχοληθούμε το θέμα της στέγασης, της ιατρικής και ψυχολογικής θεραπείας και υποστήριξης, το θέμα της ενημέρωσης σε μία γλώσσα κατανοητή για το θύμα και όλες τις άλλες μορφές συμπληρωματικής υποστήριξης και βοήθειας για τα θύματα. Απαντώντας την κυρία Ζαμπόρσκα θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί με τα θέματα πρόληψης αυτής της μάστιγας και με το θέμα της προστασίας της επανόδου και της επανένταξης αυτών των παιδιών θα, μέσα σε ένα σχέδιο δράσης για την προστασία των μη συνοδευόμενων θυμάτων. Αυτό ήταν άλλωστε ένα πολύ έντονο αίτημα της Ισπανικής Προεδρίας, κύριε Υπουργέ. Θα προτείνουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο δράση, το οποίο θα εγκριθεί τον Άνοιξη του 2010 από την Επιτροπή για να εξεταστεί κατόπιν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σχέδιο δράση θα προτείνει διάφορε λύσει για την αντιμετώπιση των κυρίων προβλημάτων <clears throat> που αφορούν τα μη συνοδευόμενα ε, ανήλικα άτομα που φτάνουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελέγει επίσης δίκιο η κυρία Ζαμπόσκα. Πρέπει να εμπλακούν και οι οικογένειες στη σε όλη αυτή τη διαδικασία φροντίζοντας περισσότερο να αποφεύγουν τα παιδιά τους τη χρήση του διαδικτύου μέσω του οποίου εκτίθενται σε νέους κινδύνους. Υπάρχει πολιτική βούληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπε και ο Υπουργός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προετοιμάσει καλά το σχέδιο οδηγίας, το οποίο θα υποβάλει σύντομα και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που με τον τρόπο αυτό μας έχει δώσει όλη του την υποστήριξη αλλά και πάρα πολύ σημαντικές κατευθύνσεις που προέκυψαν στη διάρκεια αυτής της συζήτησης τις οποίες σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές πιστεύοντας ακράδαντα ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία θα παίξει σημαντικότατο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση αυτής της φρικτής μάστιγας. Ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστώ Υπουργέ, ευχαριστώ τις δύο συγγήτριες, όλους τους ομιλητές, το προσωπικό τους ε, διερμηνείς, λύεται η συνεδρίαση.